Ε, των πολιτών. Μην το ξεχνάμε αυτό, είναι προτεραιότητα. Ευχαριστούμε. κάποιο άλλος. Κανείς. Ίσως θα μπορούσα σε τέσσερα σημεία να αναφέρω. Το πρόβλημα είναι δεδομένο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι έλαβαν λέει νέες πληροφορίες και αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Όμως δεν κατέληξαν με μια τελική θέση ακόμα. Επίσης ακούσαμε ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος εξετάζει το πρόβλημα. Όμως δεν έχουν ακόμα καταλήξει σε μια τελική θέση ή στάση από πλευράς τους. Επίσης ακούσαμε ότι δεν έχουμε ακριβή λέει, στοιχεία από τις Ιταλικές αρχές επ' αυτών τι απορρέει. Θα απομείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα παρακολουθήσουμε εκ του σύνεγγι στο τι συμβαίνει και τεκταίνεται. Θα απευθυνθούμε προς τις Ιταλικές Αρχές για να υποβληθούν περαιτέρω πληροφορίες. Επίσης θα έρθουμε σε επαφή με τους συναδέλφους μας της Επιτροπής Περιβάλλοντος, θα ζητήσουμε να μας υποβάλουν την άποψή τους επί του θέματος και επίσης προσβλέπουμε στη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση επακόλουθες πληροφορίες και θα επανέλθουμε και θα δώσουμε συνέχεια στη συνέχεια. Σας ερωτώ αν συμφωνείτε. Αν ναι, σας ευχαριστώ πολύ από πλευρά συναδέλφου μου υπενθύμησε ότι ίσως οι εκπρόσωποι από πλευράς αναφέροντος θα ήθελαν δύο λεπτά που θα χρειαζόντουσαν για να σχολιάσουν τα σχετικά. Παρακαλώ. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών που άκουσε τα αιτήματά μας, τα αιτήματα των πολιτών και τα έλαβε υπόψη της. Ελπίζουμε πολύ σύντομα τα μη χρησιμοποιηθέντα κονδύλια να χρησιμοποιηθούν επιτέλους και να επιληθεί το πρόβλημα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, κυρίε και κύριοι, προχωράμε λοιπόν. Η επόμενη αναφορά είναι η 1405 που υποβλήθηκε από έναν βούλγαρο υπήκο. Είναι ένα περίπλοκο θέμα πάλι, πάλι ένα θέμα που αφορά το περιβάλλον με επιπτώσεις στην υγεία των βουλγάρων πολιτών. Από πλευράς ε, αναφέροντος, που καθότι γνωρίζω δεν παρίσταται, και αν συμβαίνει αυτό, θα ήθελα να ζητήσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να από πλευράς δηλαδή της αντίστοιχης γενικής διεύθυνσης να μας αναφέρει ποιες είναι οι απόψεις τους. Παρακαλώ. Yeah, Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα. Εκπροσωπώ την ε, περιβάλλοντος. Δεν ξέρω αν είναι θέμα διερμηνίας. Ε, η Επιτροπή γνωστοποίησε το ότι διαδικασίες επί παραβάση σε σχέση με τη Βουλγαρία είχαν αναλυθεί για να διασφαλιστεί η ε, διαχείριση η οποία δεν προχώρησε και λόγω της υλοποίησης ε, του προγράμματος για την υιοθέτηση ενός προγράμματος αντιμετώπισης στερεών αποβλήτων όσον αφορά την περιοχή, την επικράτεια της Σόφιας. Το πρόγραμμα προβλέπει μια νέα χωματερή και την αντιμετώπιση μηχανικής ε, αντιμετώπισης ε, από πλευράς εγκατάστασης των αποβλήτων με, καθώς ξεκίνησε το 2015 αυτό οδήγησε στο να κλείσει, να κλείσει η χωματερή στο Σουχοντόι που ήταν ακριβώς αντικείμενο της αναφοράς. Το Δεκέμβριο 2012 λοιπόν μια νέα χωματερή άνοιξε όσον αφορά την οδηγία για το περιβάλλον και με το κλείσιμο των, της άλλης μονάδας. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν για την περιοχή της Σόφιας με την κομποστοποίηση ε, των ε, ουσιών για την παραγωγή με περιβαλλοντικό τρόπο της κομποστοποίησης ε, και από τον Ιανουάριο 2014 και τον Σεπτέμβριο 2015 έγιναν ε, αυτές οι εξετάσεις μετά από την εξέταση και ολοκλήρωση όσον αφορά το πρόγραμμα αυτό ε, διεπίστωσε η Επιτροπή ότι κατάφερε η Βουλγαρία να διασφαλίσει την αντιμετώπιση των υποχρεώσεών της όσον αφορά την αντιμετώπιση των στερεών αποβλήτων και έτσι έπαυσαν πλέον οι διαδικασίες ε, επί παραβάση από πλευράς της Επιτροπής. Σας ευχαριστούμε. θα ήθελα να ρωτήσω όσον αφορά τη διαδικασία επιπαραβάση. Ποια είναι η διαδικασία. Έκλεισε ή εξακολουθεί και συνεχίζεται. Η διαδικασία επιπαραβάση έχει ήδη κλείσει διότι η κατάσταση βελτιώθηκε όπως αναφέρθηκε. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων στη Σόφια πλέον και δεν υπάρχει κανένας λόγος λοιπόν σε αυτή την περίπτωση να συνεχιστεί η διαδικασία επί παραβάση. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Ερωτώ τώρα τους συναδέφους. Θα ήθελα να σχολιάσω, να παρέμβουν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αλλά έχω μια πρόσθετη ερώτηση σε σχέση με την χρήση αυτής της ε, έκτασης. Τι συμβαίνει ακριβώς εξακολουθούν να υφίστανται κίνδυνοι για το περιβάλλον εξακολουθεί να υπάρχει κάποιο έργο το οποίο γίνεται για την αποκατάσταση ή για την ε, διάθεση μιας ε, νέας έκτασης. Όχι, έκλεισε εντελώς αυτή η μονάδα και έχει ετοιμαστεί μια άλλη χωματερή και η διαδικασία αποκατάστασης συνεχίζεται. Έχει κλείσει όμως η μονάδα αυτή. Ευχαριστώ. Γιάροσλαβ, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Φαίνεται ότι οι διαδικασίες επί παραβάση έκλεισαν, μια και προς ικανοποίηση των εμπλεκόμενων μερών αυτά ε, αξιολογήθηκαν με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ Πρόεδρος. Συμφωνώ με την άποψή σας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω συμφωνεί ότι θα έπρεπε να κλείσει αυτή η υπόθεση και συνάδελφοι εξίσου Κανείς δεν είπε κάτι το διαφορετικό. Μπορούμε να κλείσουμε λοιπόν αυτή την αναφορά. Σας ευχαριστώ. Και τώρα η επόμενη αναφορά αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι 270 κάθετος 15 που έχει κατατεθεί από πλευρά του Αντρέη Καμνιεύ με συλλογή υπογραφών Πρόκειται για ένα πρόβλημα οδηγών φορτηγών επαγγελματιών αυτοκινητιστών στη Γερμανία και σε άλλες χώρες έχουν έναν ελάχιστο μισθό που, έχει, που προβλέπεται για αυτούς. Και σε σχέση με τα θέματα αυτά, τα μισθολογικά που δημιουργούν πρόβλημα, ο αναφέρον δεν παρίσταται και ερωτώ λοιπόν τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φεντερίκο Μπανκάντι ή συνάδελφο, συνάδελφο ε, ποια είναι η άποψή του να μας εκτεθούν δηλαδή απόψεις της Επιτροπής σχετικά παρακαλώ Ευχαριστώ Πρόεδρε Ουσιαστικά το πώς έχει αυτή η υπόθεση είναι ότι η διαδικασία επί παραβάση εξακολουθεί και προχωρεί έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έχει αποστείλει μια επιστολή ε, ενημερωτική σε σχέση με τις γερμανικές αρχές και με την πρόσθετη αυτή επιστολή αξιολογούμε αυτή τη στιγμή πως έχει κατάσταση και διεξάγονται συζητήσεις σε σχέση με τις γερμανικές αρχές. Όσον αφορά την ίδια την ουσία του θέματος αυτού, σε σχέση με τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά, αυτή είναι ότι χαιρετίζουμε φυσικά την εισαγωγή ενός ελάχιστου μισθού στην Γερμανία. Γενικά θεωρούμε ότι είναι ένα καλό μέτρο αυτό για να βελτιωθούν οι όροι και συνθήκες απασχόλησης και για να ε, τονωθεί ο ανταγωνισμός σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι είναι κατά μια συστηματικής υποχρέωσης επιβολής ελάχιστου μισθού σε όλες τις ε, μεταφορικές ε, ε, πτυχές, όλες τις εργασίες όσον αφορά τις μεταφορές. Υπάρχουν ίσως και θέματα περιορισμού ελευθερίας όσον αφορά παροχή υπηρεσιών και ελευθερίας κυκλοφορίας των αγαθών και γι' αυτό θα πρέπει να μην υπάρχει δυσανάλογη εφαρμογή των μέτρων αυτών από τους εμπλεκόμενους. Δεν είναι όλοι οι μεταφορείς οι οποίοι θα έπρεπε να υφίστανται σε αυτή τη ρύθμιση αυτών των διατάξεων. Αν ένας μεταφορέας για παράδειγμα διασχίζει τη χώρα χωρίς να παρέχει υπηρεσίες στην ίδια τη γερμανική επικράτεια, τότε ο οδηγός αυτού του φορτηγού δεν θα έπρεπε να απολαμβάνει τις διατάξεις του ελάχιστου αυτού μισθού όπως ισχύει για άλλες δραστηριότητες στη Γερμανία. Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι το μέτρο αυτό δεν αφορά μόνο τον ελάχιστο μισθό, αλλά οδηγεί και σε διοικητικές απαιτήσει και διοικητικές δαπάνες ε, που συνεπάγεται και σε σχέση με την γραφειοκρατική επιβάρυνση που προξενείται για μικρές επιχειρήσεις. Για όλους αυτούς τους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν πρέπει να είναι δυσανάλογη η εφαρμογή του μέτρου. Τώρα, σε ένα άλλο πλαίσιο, φυσικά οι, Ευρωπαϊ... οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενεπλάξαν στην αναθεώρηση όλου του πλαισίου νομοθετικών διατάξεων που διέπουν τις μεταφορές και των κοινωνικών κανόνων που αφορούν τις μεταφορές. Σε σχέση με την αναθεώρηση λοιπόν και της απόσπασης εργαζομένων που ισχύει για όλους τους τομείς και για τις μεταφορές, θεωρούμε ότι στο επίπεδο των υπηρεσιών μπορεί να υπάρχουν πιθανώς ευκαιρίες με την αναθεώρηση της κοινωνικής νομοθεσίας και διατάξεων να αποσαφινιστεί σε ποιο εύρος η απόσπαση εργαζομένων θα ίσχυε όσον αφορά τον τομέα των μεταφορών. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διαχωριστεί απόλυτα σε σχέση με την περίπτωση αυτή στην Γερμανία και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις για παράδειγμα που αφορούν τη Γαλλία <clears throat> και πιθανώς και άλλα κράτη-μέλη σχετικά. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ. Και θα ήθελα να δώσω τώρα τον λόγο στους συναδέλφους να παρέμβουν. Ρόσλα. Και μετά ίσως κάποιος άλλος συνάδελφος. Μια και κάνουμε λόγο για πολυ, πολωνική αναφορά, πάρτε εσείς πρώτος τον λόγο, παρακαλώ. Ε, Εντάξει, ευχαριστώ. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο θα είχα, μια και συνεχίζονται οι διαδικασίες και δεν έχει ακόμα διευθετηθεί το θέμα. Θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Αυτό είναι το μόνο σχόλιο που έχω σε αυτή τη φάση. Πρόεδρος, πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Εσείς, ευχαριστώ πρόεδρε. Από την Επιτροπή Μεταφορών που πραγματικά θα θέλαμε να δούμε ποιες, θα είναι, είναι οι εξελίξεις σχετικά και στρεφόμαστε και προς την Επιτροπή αυτή τη στιγμή σε αυτή τη φάση διότι ήδη αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και είδαμε εντωμεταξύ ότι και κάποια άλλη δύο κρατημέλη για παράδειγμα, έχουν κατά κάποιο λόγο εισαγάγει παρόμοια συναφή μέτρα. Γαλλία για παράδειγμα και κάποιο άλλο κράτος που προετοιμάζουν αντίστοιχα μέτρα. Και κάθε χώρα φυσικά έχει το δικαίωμα να αποφασίζει πόσα ισχύει ο ελάχιστος μισός. αυτό δεν είναι το ζήτημα. Συμφωνούμε επ' αυτού. Ιδιαίτερα όμως όταν εξετάζει κανείς τον τομέα των μεταφορών, τις μεταφορικές εταιρείες και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες εταιρείες από πλευράς των μεταφορών υπάρχει ιδιαίτερη επιβάρυνση για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ικανοποιήσουν όλες τις διαφορετικές απαιτήσει με τις διατάξεις που εισάγει η Εθνική Νομοθεσία για αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και φυσικά σε σχέση και με την, ε, τον διαχωρισμό ή την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έλεγα και σε σχέση ακόμα και με την ε, οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων, ουσιαστικά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε με μεγαλύτερη σαφήνεια τι συμβαίνει και να δούμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις προτάσεις αυτές για την απόσπαση εργαζομένων. Πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να λάβουμε κάποια, να τοποθετηθούμε σχετικά για τη Γερμανία ή άλλες χώρες. Χωρίς να προωθείται η διαδικασία επί ε, παραβάση, μπορούμε να πούμε ότι δεν ε, βρίσκεται η λύση η θα έπρεπε να επιλεγεί. Ευχαριστώ πολύ. Εσείς έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ε, Σας ευχαριστώ. Είναι δύσκολο το έργο αυτό. Είναι δύσκολο γιατί εμπλέκονται πολλά θέματα και ερωτήματα τα οποία πρέπει να τεθούν και να απαντηθούν. Όταν εισήχθησαν ή όταν εισάγονται τέτοια μέτρα. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις που θα μπορούσαν να έχουν σε επιχειρήσεις, σε πύχη της Πολωνίας, διότι στο τέλος τέλος υπάρχουν υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και αυτό τις επιβαρύνει ιδιαίτερα. Και θα πρέπει να δούμε επίσης και το θέμα της απασχόλησης στον τομέα αυτό, για παράδειγμα των επαγγελματιών οδηγών στις ε, μεταφορές και την κατάστασή τους. Σημαντικό θα ήταν λοιπόν να δούμε τις επιπτώσεις ε, που θα υπάρχουν. Επιπτώσεις ε, και για τις επιμέρους χώρες ξεχωριστά. Φυσικά είναι χαμηλότερος ο μισθός σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες εναντί άλλων. Όμως δεν είναι απλό το θέμα να πει κανείς ότι θα χαιρόντουσαν οι οδηγοί απλά και μόνο με μια διάταξη που μπορεί, θα μπορούσε ίσως να διασφαλίζει ε, έναν μεγαλύτερο μισθό διότι το θέμα είναι ποιες άλλες συνθήκες θα ισχύουν και ποιες επιπτώσεις θα υπάρχουν στους όρους απασχόλησης για αυτές τις επιχειρήσεις. Στο τέλος τέλος θα υπάρξουν ίσως και απολύσεις από κάποιες επιχειρήσεις και θα πρέπει να ζητήσουμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι ότου υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα. Να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις, πώς μπορούν αυτές να εκτιμηθούν. Χρειαζόμαστε όμως γι' αυτό μια, ένα αρκετά υψηλό ε, βαθμό πιθανότητων για να ισχύσει και να μπορέσει να λειτουργήσει. Έχω πει πολλές φορές ε, και στην Επιτροπή μας ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία με την Επιτροπή Απασχόλησης. Ε, εδώ και δύο χρόνια ασχολούμαστε στην Επιτροπή Απασχόλησης για το θέμα και περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα ε, της διαδικασίας αυτής επί παραβάση. Επίσης υπάρχει το πρόβλημα το τι καθεστώς έχει η εταιρεία αυτή μεταφορική. Υπάρχουν πολλά σημεία, πολλές πτυχές. Εγώ εκπροσωπώ τη Λετωνία ένα κράτος Ανατολικής Ευρώπης και σίγουρα έχουμε και εμείς προβλήματα με τους ε, δικούς μας οδηγούς φορτηγών και τις διάφορες εταιρείε. Θα πρότεινα φυσικά να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Θα έχουμε βέβαια και ένα νέο δίκτυο πώς λεγόταν το ξέχασα, αλλά τέλος πάντων θα έχουμε ένα δίκτυο συνεργασίας ε, μεταξύ επιτροπών. Petition Network, α ναι, το δίκτυο αναφορών. Εγώ εκπροσωπώ την Επιτροπή Απασχόλησης σε αυτό το δίκτυο, τέλος πάντων. Ε, εγώ θα ήθελα να το υποβάλω υπόψη, να το θέσω. Μήπως θα μπορούσαμε να το συναντήσουμε το δίκτυο δεν πώς θα δημιουργηθεί, πώς θα συσταθεί αυτό το δίκτυο, αλλά θα πρέπει ίσως να το συζητήσει αυτό το θέμα. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Στρέφομαι προς τους συναδέλφους. Έχετε να προσθέσετε κάτι ακόμη, αν όχι. Αν όχι, λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να συνοψίσουμε το πράγμα ως εξής επιτεύχθη ο πρώτος στόχος, δηλαδή πλέον το πρόβλημα έγινε γνωστό, το έχουμε αντιληφθεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ε, ότι πρέπει τώρα να το επιλύσει. Θεωρώ ότι καλό είναι να μείνει ανοιχτή αναφορά. Η Κομισιόν έχει σωστή στάση, προσπαθεί να βρει ε, τρόπο να λύσει το πρόβλημα. Επίσης χαίρομαι που ασχολούνται και οι άλλε δύο ε, του Κοινοβουλίου από διαφορετική οπτική γωνία καθεμία ασχολούνται με το θέμα αυτό. Άρα συμφωνώ με τους συναδέλφου ότι θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα αναμένουμε τις ε, μελλοντικέ εξελίξεις. Ευχαριστώ. Και τώρα κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναφορά που έχουμε στην ημερήσια διάταξη είναι 804 του 2015 από Ιταλό υπήκο για την υγειονομική περίθαλψη σε Γερμανία και Ισπανία. Το βλέπω στα έγγραφά μου δεν είναι εδώ ο αναφέρον. Όμως, μας έχει υποβάλει γραπτό στην θέση του και την έχουμε μελετήσει. Μαρία Λουίζα, Βαντέσκεν ή κάπως έτσι. Ε, θέλετε παρακαλώ να μας πείτε την άποψη της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα αναφέροντα έλεγε ότι υποθέτει ότι είναι ασφαλισμένο στην χώρα καταγωγής του ο εν λόγω αναφέρον. Άρα θα έπρεπε να έχει αυτό το έγγραφο S1, με βάση το οποίο δικαιούται η υγειονομική περίθαλψη στο κράτος μέλος το οποίο διαμένει. Το πρόσφατο μήνυμα όμως ε, του αναφέροντα μεταφέρει δύο στοιχεία σημαντικά τα οποία δεν γνωρίζαμε. Πρώτον, ότι δεν πληρώνει πλέον εισφορά στην Ιταλία, δεν είναι ασφαλισμένο πλέον στην Ιταλία. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι δεν πληρώνει και τι φορέ κοινωνική ασφάλιση στην Ισπανία. Ούτε εκεί. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κανονισμοί συντονισμού. Δεν μπορεί να χορτέψει ε, οικονομικά. Το πρόβλημα είναι ότι ο συντονισμό, αυτό, αυτός ο μηχανισμός Το 888 και 989-2007 ουσιαστικά συντονίζουν, όπως λέει και το όνομά τους, ε, δεν εναρμονίζουν τα πράγματα, οπότε το κάθε κράτος μέλος μπορεί να ορίσει τις προποθέσεις ε, και τα πιο αναλυτικά ε, στοιχεία των ασφαλιστικών συστημάτων. Στην Ισπανία δηλαδή. Ισχύει ακριβώς το ίδιο. Η Ισπανία είναι ελεύθερη να αποφασίσει πώς κάποιος θα προσχωρεί και θα εγγράφεται στο ασφαλιστικό σύστημα. Επειδή υπάρχουν διαφορετικά διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών και των ασφαλιστικών συστημάτων που δεν υπερπηδούνται από αυτό το μηχανισμό συντονισμού ή μεταφορά το ένα κράτο στο άλλο δημιουργεί ζητήματα. Πρώτον, στα δικαιώματα, ε, στις παροχές και στις εισφορές ε, κοινωνική ασφάλισης. Για ανενεργά οικονομικά άτομα, η χώρα καταγωγής είναι η χώρα ασφάλισης η ε, χώρα κατοικία, συγγνώμη, που σημαίνει ότι στην Ισπανία πρέπει να ασφαλιστεί ο εν λόγω υπήκος. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την οδηγία 38 του 2004 για το δικαίωμα των ε, πολιτών της Ένωσης και των μέλων της οικογένειά τους να μπορούν να διαμένουν ε, ελεύθερα ε, στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Υπάρχει το άρθρο 7 συγκεκριμένα, το οποίο θεσπίζει προϋποθέσεις ε, για την νόμιμη έδρα ενός κατοίκου που μετακινείται σε ένα άλλο κράτος μέλος για ανενεργά οικονομικός άτομα. Δύο είναι οι προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι να έχουν επαρκείς πόρους στη διάθεσή τους και για τα μέλη της οικογένειας ώστε να μην αποτελούν βάρος ε, για το κοινωνικό σύστημα ασφάλισης της χώρας ε, στην οποία ε, κατοικούν πλέον. Και το δεύτερο και σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να έχουν μια συνολική ασφαλιστική κάλυψη σε αυτό το κράτος, το οποίο πλέον διαμένουν. Υπήρχε ξεπρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου ε, εναντίον Ηνωμένου Βασίλειου Βασιλείου 2014 που μιλάει για αυτή την προϋπόθεση για τη χορήγηση κοινωνικών επιδομάτων, δηλαδή των ασφαλισμένο στη χώρα ε, διαμονή ένα ε, ε, πολίτη τη Ένωση. Με βάση όλα αυτά λοιπόν θεωρούμε ότι ο αναφέρον θα πρέπει να γραφτεί στο σύστημα ασφάλισης τη χώρα, στην οποία κατοικεί, δηλαδή στην Ισπανία και θα πρέπει εκεί να τηρεί τι ίδιε υποχρεώσει με του υπόλοιπου ασφαλισμένου στην Ισπανία, οι οποίοι φυσικά βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με αυτόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Καλά κατάλαβα όμως τη θέση σας. Ούτε η Γερμανία δηλαδή, ούτε η Ισπανία παραβιάζουν ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία με τις πρακτικές τους που έχουν σε ισχύ. Έτσι είναι τα πράγματα, απάντηση. Από τα γεγονότα ε, που παρουσίασα αναφέρουν, λέμε ότι για οικονομικά ανενεργά άτομα αυτός ο υπήκος θα έπρεπε να είναι εγγεγραμμένος ε, στην, ε, στο Ισπανικό ασφαλιστικό σύστημα. Η Ισπανία δεν παραβίασε την προκειμένη περίπτωση την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ κυρία Πέτερα. Ευχαριστώ. λείπουν κάποιες πληροφορίες. Μας στάθηκαν πληροφορίες, αλλά θα πρέπει να δούμε αν έγινε η προσπάθεια, αν καταβλήθηκε η προσπάθεια, τα δικαιώματα του αναφέρω να τα διασφαλίσει στη χώρα όπου έχει την, στην οποία κατοικεί. Δεν γνωρίζουμε ποιος εξέδωσε αυτή την κάρτα ασφάλισης ασθένειας και εδώ τίθενται θέματα και δεν γνωρίζουμε αν στράφηκε στην ε, ε, αρμόδια υπηρεσία ή ανέθεσε έτοιμα ώστε να εκδοθεί μια τέτοια κάρτα ασφάλισης. Πρέπει να αποσαφινιστούν αυτά. Πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Θα ήθελα όμω να στραφούμε στον αναφερόμενο και να ζητήσουμε για ε, να δοθούν πρόσθετες πληροφορίες και αποσαφινίσεις. Sorry, be a technical problem. There is no English interpretation. πρόβλημα και δεν υπήρχε αγγλική μετάφραση. Τώρα είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Ωραία. Άρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Ο Λαβ. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω με αυτό που είπε η Γιούλια. Αλλά να πω ίσως το ανάποδο θα μπορούσαμε να κάνουμε, να καταρτήσουμε μια επιστολή για τον αναφέροντα, όπου θα του ζητούμε να μας απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Δηλαδή πριν μας στείλει την αναφορά σε τι ενέργειες προέβη. Μπορούσε ή δεν μπορούσε να λάβει γνώση των κοινωνικών επιδομάτων ε, ή των άλλων παροχών υγείας στη χώρα κατοικίας του και μέχρι να λάβουμε την απάντηση θα μπορούσαμε ήταν να διατηρήσουμε μετά, δηλαδή αφού πάρουμε την απάντηση να δούμε αν θα κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά ή να την κλείσουμε πάντα με βάση τα μας απαντήσει αναφέρουν. Η κυρία Σντανόκα. Ευχαριστώ. Έχω μία ερώτηση προς την εκπρόσωπο της Κομισιόν. Δεν κατάλαβα. Ε, το σημείο της δήλωσής σας όπου λέγατε κάτι για την κατοικία. Υπάρχει ένα θέμα ε, που το αντιμετωπίζουμε ποια είναι η συνήθις ε, διαμονή, συνήθις τόπος διαμονής, κατοικία. Ε, δεν είναι σαφές αυτό και δεν κατάλαβα εσείς που αναφερόσασταν ακριβώς. Να απαντήσω, λέει εκπρόσωπος Κομισιόν. Ναι. Επειδή δεν είχα αγγλική μετάφραση, δεν άκουσα τι είπε η συνάδελφος ε, η κυρία. Θα απαντήσω στα άλλα ερωτήματα. Εγώ μιλούσα για το legal residence test υπάρχει η οδηγία για την ελεύθερη μετακίνηση προσώπων. Όταν μιλάμε για συνήθι τόπο διαμονή, habitual residence, αυτό ο όρο ε, είναι σε αυτού του κανονισμού συντονισμού, που σημαίνει που είναι το κέντρο των ενδιαφερόντων κάποιου προσώπου. Και με βάση αυτό αποφασίζονται τα επιδόματα στα οποία ε, έχει δικαίωμα. Η οδηγία περί ελεύθερης κυκλοφορίας, όταν μιλάμε για ε, τον νόμιμο τόπο, νομικό τόπο διαμονής, εγώ μιλούσα για αυτά τα ανενεργά άτομα. Για να μπορούν να κατοικούν ε, νομίμως ένα κράτος μέλος, θα πρέπει να εκπληρούν δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι να έχουν επαρκείς πόρους οικονομικούς για να μην επιβαρύνουν τα ασφαλιστικά συστήματα, κοινωνικά συστήματα στη χώρα που διαμένουν και δεύτερον να έχουν και μία πλήρη κάλυψη ασθενείας, να έχουν ασφάλιση ασθενείας. Ευχαριστώ. Ελπίζω να είναι σαφές τώρα. Η κυρία Σντανόκα. Εγώ βλέπω εδώ ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ε, σε ό,τι αφορά τους ορισμούς. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβείς οι, αρισμοί, οι ορισμοί και νομίζω ότι γι' αυτό ακριβώς έχουμε πρόβλημα. Εκκρέμει αυτό το ζήτημα τι είναι συνήθις τόπος διαμονής και οι σχετικοί ορισμοί, οι συναφείς αν δηλαδή κάποιος πολίτης μπορεί να διαμένει ουσιαστικά σε δύο ή περισσότερα κράτη-μέλη. κομισιών. Στου κανονισμού συντονισμού ορίζεται αυτό το συνηθιστό διαμονή και στον εφαρμοστικό κανονισμό. Επίσης υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων οι εθνικές αρχές μπορούν ε, να διακριβώσουν που έχει κάποιος ε, τη συνήθεια του διαμονή και για τους φοιτητέ, για παράδειγμα, είναι η χώρα από την οποία προέρχεται, προέρχονται τα έσοδα του, το εισόδημα του φοιτητή. Πρόεδρος. Εγώ θυμάμαι την πρώτη πρόταση της κυρίας που είπε ότι υπάρχει συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά είπατε ότι δεν έχει λύθει το πρόβλημα, αν κατάλαβα καλά. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια νομικά δεσμευτική αναλυτική λύση στο πρόβλημα. Και ίσως τελικά το πρόβλημα βρίσκεται ακριβώ σε αυτή την γκρίζα ζώνη. Για να είμαι ειλικρινή, εγώ θα πρότεινα με βάση τη δήλωση της Κομισιόν να κλείσουμε την αναφορά. Άκουσα όμως ε, τα διλήμματα που έχουν συνάδελφοι. Οπότε τώρα τίνω κι εγώ, όπως ανέφερε ο Γιάροσλαβ, τίνω κι εγώ να προτείνω να ζητήσουμε από τον αναφέροντα να μας δώσει ακόμα πιο αναλυτικές πληροφορίες συγκεκριμένα για το τι ενέργειες έκανε, επειδή δεν έχουμε καμία σχετική πληροφορία. Και με βάση αυτές τις πληροφορίες έπειτα να ξαναδούμε το ζήτημα και να αποφασίσουμε κατά πόσον θα την κλείσουμε, θα την αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Προ το παρόν όμω δεν έχουμε επαρκεί πληροφορίε στη διάθεσή μα. Σε σχέση, επαναλαμβάνω, με τι ενέργειε στις οποίες προέβη ο εν λόγω υπήκο. Ε, δέχεστε την αποψή μου, συνάδελφοι. Αν ναι, περνάμε στην τελευταία για σήμερα αναφορά. Είναι υπαριθμόν 0789 ε, κάθετος 2015 από έναν Λευκορώσο πίκο που ζει και στο Βέλγιο όμως. Λέγεται Αντρέι Σουμάρ. Και η αναφορά αυτή αφορά πολωνική θεώρηση διαβατηρίου. Θεωρεί ότι γίνονται κάποια περίεργα πράγματα στη Λευκορωσία, αναφέρουν. Έχουμε τον αναφέροντα εδώ. Θα του δώσω τώρα το λόγο. Και θα τον παρακαλέσω να μας παρουσιάσει μέσα σε πέντε λεπτά την υπόθεση του. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Ε, dear sirs, madams, in July Τον Ιούλιο του 2015 υπέβαλα μία αναφορά για το λαθρεμπόριο ε, πολωνικών θεωρήσεων ε, την υπέβαλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εν συνεχεία, ε, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι, μπορούμε να πούμε ότι αναφορά αυτή αφορά την απειλή της τρομοκρατίας. Στα τελωνία πληρώνουμε 400 ή 500 ευρώ σε ενδιάμεσους. Ε, δεν χρειάζεται κανένας για να πάρει ε, πολωνική θεώρηση να πάει στο προξενείο. Η Ευρώπη αξίζει 400 ή 500 ευρώ. Ε, με 400 ευρώ, ας πούμε, ε, μπορεί να γίνει μία τραγωδία. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους οι οποίοι κατ' επανάληψη κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι υποτροπιάζοντες εγκληματίες. Η... Αυτό ξεκίνησε το 2011 ε, πολλοί ξένοι κρατήθηκαν ε, γιατί έκαναν αυτή τη δουλειά και δεν τους επιτρέψαμε να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά παρόλα αυτά είχαν θεωρήσεις πολωνικές. Τα... Στη Λευκορωσία ε, οργανώσαμε... Συγγνώμη, μάλλον δεν υπάρχει κανένα ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ερευνά αυτά τα εγκλήματα για τις απάτες των θεωρήσεων. Νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να γίνει κάποια έρευνα. Να σα επιστήσω την προσοχή ότι με βάση τις πληροφορίες που έλαβα από τη γραμματεία της Επιτροπής ΠΕΤΗ, οι πολωνικέ αρχές δεν απάντησαν στο ερώτημα που τους ε, υποβάλαμε και δεν σχολίασαν την αναφορά. Οι πολωνικές αρχές θα πρέπει, προσπαθούν μάλλον να αποφύγουν τις ευθύνες τους. Γιατί μπορεί η απάντηση αυτή να χρησιμοποιηθεί αντίον τους. Σας καλώ να μην πάρει τις ευθύνες για εγκλήματα που κάνουν άλλοι. Πρόσφατα έχουμε λάβει προειδοποίησεις για πιθανές τρομοκρατικές επιθέσεις. Από εδώ και πέρα, μετά από κάθε τέτοια προειδοποίηση, κάθε από εσά θα πρέπει να κρατάει την ανάσα του και να προσεύχεται ότι οι τρομοκράτες δεν θα έχουν και να ελπίζουν ότι θα έχουν μία ε, θεώρηση Σέγγεν. Αλλά εάν ο τρομοκράτης έχει τέτοια θεώρηση Σέγγεν, καθένας από εσά θα αισθάνεται ένοχος και θα ε, ε ποτέ τον εαυτό του. Ε, το κίνημα αυτό Renaissance ξεκίνησε τις έρευνες για τις παράνομες θεωρήσεις στη Λευκορωσία το 2012. Μετά από ένα χρόνο οι τοπικές αρχές άρχισαν να ασκούν πίεση σε εμά. Χρειάστηκε να κλείσουμε δύο ιστοσελίδες, του κινήματος Renaissance και να μειώσουμε στον ελάχιστο βαθμό τις δραστηριότητε μας. Μετά από ένα χρόνο χρειάστηκε να φύγω από τη Λευκορωσία, αναγκάστηκα να φύγω. Οι απαταιώνε που είχαν οργανώσει αυτή, αυτό το λαθρεμπόριο με τι θεωρήσει στη Λευκορωσία είχαν ε, βρει πολύ, ένα θαυμάσια, μια θαυμάσια ας πούμε, δουλειά σε αυτή τη χώρα, γιατί το καθεστώ τη Λευκορωσία δεν προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών ε, για να υποβάλουν ε, χαρτιά και να λαμβάνουν τι θεωρήσει έγκαιρ. Εγώ έκανα έκκληση στις αρχές της Πολωνίας ε, και του ζήτησα άσυλο. Ε, ξόδεψα ένα χρόνο σε πολωνικά στρατόπεδα ε, προσφύγων. Ε, υπέβαλα διάφορες προσφυγές, ε, μίλησα για αυτή την απάτη για τις θεωρήσεις ε, και όμως δεν έγινε τίποτα. Είναι σαφές ότι το πολωνικό νομικό σύστημα είναι ατελές για να μην πω διεφθαρμένο. Ε, ασκείται απίστευτη πίεση και σε μένα όταν ήμουν στην Πολωνία αλλά και σε άλλους. έλαβα απειλές και χρειάστηκε ε, να προσέξω και γιατί μου επιτέθηκαν διάφοροι και όταν, ε, όταν έφυγα για το Βέλγιο το 2015 πονούσαν οι γροθιές μου από τις ε, γροθιές που αντάλλασα με διάφορους. Ε, δυστυχώς όλα αυτά ε, γίνονται, ξανάρχισαν όλα αυτά τα προβλήματα που είχα ξανάρχισαν στο Βέλγιο. Ε, Έχω περάσει και ένα χρόνο εδώ στο στρατόπεδο προσφύγων, στο Βέλγιο δηλαδή. Ε, μιλάμε για φοβερή πίεση, ε, μιλάμε για επιθέσεις, για δηλητηρίαση του φαγητού μου και όλα αυτά. Χρησιμοποιήθηκαν εναντίον μου. Έχω στείλει επιστολές ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάποιος προσπαθεί να με σταματήσει για να μην δημοσιοποιήσω αυτή την ε, ιστορία για τις παράνομες θεωρήσεις του Σέγγεν. Ποιος το κάνει αυτό. Θέλω να επιστρέψω τον ετών δυνατόν στην ε, χώρα μου. Δεν έχω δει του γονεί μου εδώ και δύο χρόνια, αλλά δεν μπορώ να επιστρέψω γιατί είμαι ο μοναδικός ε, που ζητάει να ερευνηθεί αυτή η απάτη για τις θεωρήσεις. Το ζητάω από τι αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω μετά από αυτή τη συνάντηση να με υποστηρίξετε και ελπίζω να σταματήσουν οι απειλέ εναντίον μου. Σα ευχαριστώ. <clears throat> Ευχαριστώ. Κύριε Σουμαρού, Σουμάρ, σας δώσαμε την ευκαιρία να μιλήσετε για το πρόβλημα. Δημοσιοποιήθηκε το θέμα που θέλατε. Θα ήθελα να διαιρέσουμε το θέμα αυτό σε δύο υποσημεία. Καταρχάς, δεχθήκατε κάποιες επιθέσεις, μας είπατε εσείς. Φυσικά τις καταδικάζουμε, προφανώς. Σας διαβεβαιώ ότι έχετε την απόλυτη συμπαστασή μας. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι το σημείο που υπογραμμίζετε στην αναφορά σας, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λέτε ότι αν πληρώσει κανείς 400 και 500 ευρώ μπορεί να πάρει μια θεώρηση Σέγγεν και χάρη σε αυτή μπαίνει στο Σέγγεν. Έχετε, δηλαδή υπονοείτε ότι οι διπλωμάτες της πολωνικής δημοκρατίας εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρή κατηγορία, σοβαρότατος ισχυρισμό και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Είναι εδώ παρόν ο εκπρόσωπος της μόνιμης ε, πολωνικής αντιπροσωπείας. Θα ήθελα να του δώσω το λόγο, που είναι μια κυρία. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ στην κατηγορία διάπραξης αυτού του εγκλήματος όπως αναφέρεται από τον αναφερόμενο. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Πολωνίας από πλευράς του Προέδρου του Ιδρύματος Ρενεσάνς Αναγέννησης έλαβε επανειλημμένα ε, αναφορές για αυτές τις ε, για αυτή την υπόθεση με επίκληση ε, διάπραξης ε, εγκλημάτων και ότι συμπράττουν κάποιοι στην διάπραξη αυτών των εγκλημάτων. Και σε σχέση με το ανώτατο δικαστήριο και την εξέταση καταδείχθηκε ότι πρόκειται για ένα σύστημα ηλεκτρονικών επικοινωνιών εκτός ε, δικτύου και ότι δεν υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά το πολωνικό προξενείο και μετά από τις αντίστοιχες εξεταστικές ενέργειες σε αρκετά μέρη και κατά τη διάρκεια αρκετών μηνών έγιναν διακριβωτικές ενέργειες και στην πρεσβεία στο Μίνσκ και τον Νοέμβριο 2013 κανένας από τους ελέγχους δεν κατέδειξε ότι συνέβαιναν τέτοιου είδους ε, γεγονότα και ότι υπάρχει πραγματικά το βάσιμο τέτοιων κατηγοριών. Πρόκειται λοιπόν σε σχέση με την κατάθεση κάποιας αίτησης ή ε, αιτήματο ε, στο προξενείο, σε προξενείο, υπάρχει και μια ε, υπηρεσία διαμεσολάβησης, όμως δεν υπάρχουν κάποια τεκμήρια από πλευράς του κυρίου Σούμαρ που να αποδεικνύει κάτι το οποίο από αυτά τα οποία επικαλείται. Και το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει καμιά σχέση λοιπόν και καμιά εμπλοκή με όλα αυτά. Και όσον αφορά τώρα τους πολίτες της Λευκορωσίας που μπορούν και θέτουν αιτήσει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, υπάρχει και μια συμφωνία συνεργασίας από πλευράς πολωνικής κυβέρνησης για την ε, προώθηση τέτοιου είδους ε, θεωρήσεων. Πρόκειται για οκτώ κέντρα θεωρήσεων διαβατηρίων όπου είναι δυνατόν να τεθούν αιτήσει και να εκδοθούν τέτοιου είδους ε, θεωρήσεις όταν υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ε, που συνενώνονται. Τώρα, σε σχέση με την ε, εμπλοκή του Υπουργείου Εξωτερικών αυτή είναι ανύπαρκτη, δεν είναι δεδομένη σε σχέση με αυτές τις ε, κατηγορίες που γύρονται. Και πρόκειται και για ηλεκτρονικά μέσα, γίνεται κάθε προσπάθεια ώστε από πλευράς της διοίκησης ε, να γίνονται όλα εύθετα. Και τώρα, για παράδειγμα, όταν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις ε, και με προγράμματα και προθεσμίες που δίνουν την δυνατότητα σε κάποιους άμεσα να παρέμβουν και να δημιουργήσουν κάποια ηλεκτρονικά προβλήματα. Εδώ λοιπόν σε σχέση με την αλλαγή των προθεσμιών που ήταν μια προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά, μέσα στο πλαίσιο του συστήματος που ακολουθείτε, πρέπει λοιπόν να υπάρξει τροποποίηση κάποιων διαδικασιών εφόσον κάποια πράγματα δεν λειτουργούν και θα υπάρξουν και περαιτέρω ρήτρες ασφα... δικλείδες ασφαλείας ώστε να μπορέσουν τα πράγματα να λειτουργούν, να μπορέσουν να λειτουργήσουν χωρίς προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε ότι μπορούν να διευκολύνουν αυτές, αυτές οι τροποποιήσεις και ένα θέμα τώρα που αφορά τις ε, ε, διαδικασίες μεταξύ των δυνατοτήτων αριθμού θεωρήσεων που εκδίδονται σε σχέση με τις αιτήσει που κατατίθενται και να δούμε το ποσοστό το οποίο ε, καλύπτει με επιτυχία τις θεωρήσεις αυτές. Πρόκειται και για μια κατά τα άλλα επιβάρυνση και μέσα από χίλια, ε, χίλιες αιτήσει που τίθενται κατατίθενται υπάρχει ένα μικρό ποσοστό, υπάρχουν λίγοι, λίγες θέσεις, λίγα στελέχη ε, που ε, ε, διευκολύνουν. Υπάρχουν λοιπόν τεχνικά προβλήματα τα οποία αναφύονται και ζητήθηκε από τις πολωνικές αρχές να αλλάξει αυτή η κατάσταση, ωστόσο δεν άλλαξε τίποτα και πήραμε αρνητικές τοποθετήσεις σε σχέση με τις, ε, τους Λευκορώσους. Αν δεν αλλάζει λοιπόν τίποτα από αυτά, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι δυνατόν όλοι να μπορούν να θέτουν αιτήσει όπως το... I Σας ευχαριστούμε. Ε, Μπορώ να ρωτήσω για κάποια λίγα λεπτά σε σχέση με την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να την ακούσουμε και εσείς θα είσαστε ο τελευταίος που θα ε, παρέμβει. Λοιπόν, να ζητήσουμε λοιπόν από τον εκπρόσωπο την Ευρωπαϊκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Γκαμπριέλα Σμίτ ή ε, Λίμαν Σάξ, να μας εκθέσουν τις θέσεις της Επιτροπής. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ομιλώ εξ ονόματος της Επιτροπής. Η Επιτροπή έλαβε αρκετές, έλαβε πολλά παράπονα από τον κύριο Άντρε Σούμαρ για το θέμα της ε, εικαζόμενης ύπαρξης ενός εγκληματικού δικτύου που ε, καταχρηστικά εκμεταλλεύεται τις θεωρήσεις διαβατηρίων στην Λευκορωσία. Είχαμε και εννέα επιστολές ε, σε σχέση με τον πρόεδρο της Επιτροπής Jean-Claude Juncker την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας Φεντερίκα Μογκερίνη, δύο επιστολές προς τον Επίτροπο Αβραμόπουλο, υπεύθυνο για θέματα μετανάστευσης και επίσης ε, ε, λήφθηκε μια επιστολή προς τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής κύριο Τίμερμανς. Ωστόσο δεν έτυχε απάντηση επειδή ε, ε κατέφθασε με καθυστέρηση. Ο αναφέρον ισχυρίζεται ότι υπάρχει ένα εγκληματικό δίκτυο το οποίο εκμεταλλεύεται τις θεωρήσεις διαβατηρίων, θεωρήσεις ε, Ωστόσο δεν μπόρεσε να αποδείξει την ύπαρξη ενός ε, τέτοιου ε, δικτύου, εγκληματικού δικτύου. Από τα στοιχεία που αναφέρονται σε σχέση με την αλληλογραφία, μόνο ένα υπάρχει μόνο μία παρατυπία που διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αληθεύει. Σε σχέση με την πρόσβαση δηλαδή στις ε, ηλεκτρονικές καταχωρήσεις ε, και εκδόσεις ε, θεωρήσεων σε σχέση με τη Λευκορωσία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήρθε συνέχεια σε επαφή με τις προξενικές πολωνικές αρχές και το Πολωνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και αυτό που διακριβώσαμε ήταν από πλευράς μας ότι η Πολωνία είχε λάβει και ελάμβανε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διαθετηθεί αυτή η κατάσταση και σε σχέση και με τον εκπρόσωπο της μόνιμης πολωνικής αντιπροσωπείας αυτό διασφαλίστηκε. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν βρήκε να υφίσταται κάποια παραβίαση ή παράβαση ευρωπαϊκής νομοθεσίας από πλευράς της Πολωνίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε σχέση με τις ε, θεωρήσεις όσον αφορά τη Λευκορωσία είχαν εκδοθεί σε σχέση με τα όσα προβλεπόντουσαν με τον κανονισμό 810-2009 δώσαμε στη συνέχεια πέντε απαντήσεις στον αναφέροντα. Δηλαδή 17 Δεκεμβρίου 2015 όπου λεπτός τον ενημερώσαμε ότι δεν βρέθηκε καμιά παρατυπία όσον αφορά την ύπαρξη κάποιας α, ε, καταχρηστικής πρακτικής α, ε, ε, όσον αφορά την έκδοση θεωρήσεων όσον αφορά τη Λευκορωσία από πλευράς Πολωνίας. Και μετά με επιστολή τη, κατά την 26 Ιανουαρίου 2016 επαληθεύθηκε ότι η απάντηση είχε αποσταλεί επιβεβαιώνοντας την προηγούμενη τοποθέτηση. Μετά τον Φεβρουάριο 2016 με τρίτη επιστολή επιβεβαιώνεται ήδη για άλλη μια φορά η απάντηση που είχε δοθεί σε σχέση με τα θέματα που επανειλημμένα είχαν τεθεί από τον αναφέροντα. Επιβεβαιώθηκε λοιπόν η τοποθέτησή μας στις 18 Μαρτίου 2016, σύμφωνα με τον κώδικα χρηστών ε, αρχών διαχείρισης και διακυβέρνησης όσον αφορά το κοινό, ενημερώθηκε και πάλι ο αναφέρον ότι αποφάσισε να μην δώσει συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση, μια και δεν κατατέθηκαν, δεν συνελέγησαν νέα ε, στοιχεία όσον αφορά την ύπαρξη ενός τέτοιου δικτύου ή τα όσα ε, ισχυριζόταν ο αναφερόμενος. Μια και υπήρχε πυκνή αλληλογραφία από πλευρά του κυρίου ε, Σούγα από πλευράς της ε, υπηρεσίας για θέματα μετανάστευσης υπήρξε απάντηση που απεστάλλει ε, επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά τις τοποθετήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα θέματα αυτά μέσω της αλληλογραφίας που είχαμε με τον αναφέροντα. Θέλω να αναφέρω ότι εξετάστηκαν τα θέματα αυτά ιδιαίτερα όσον αφορά το προβληματικό θέμα της, ε, ε, των ε, αιτήσεων καταχωρήσεων και εκδόσεων διαβατήριων μέσω των κέντρων θεωρήσεων όπως αποκαλούνται έχουν ε, τροποποιηθεί τα πράγματα, μπορούν περισσότερες ε, αιτήσει να τεθούν μέσα σε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα ως διορία και να διευθετηθούν. Και αν υπήρχε οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα την οποία θα μπορούσαμε να, να ανοιχνεύσουμε θα ήταν έργο και πράξεις ε, πολιτών της Λευκορωσίας ε, που θα παρενέβαιναν ε, ώστε να προσπαθήσουν να πωλήσουν τέτοιου είδους υπηρεσίες μέσω τέτοιων θεωρήσεων. Ωστόσο δεν υπήρχε καμία εμπλοκή πολωνικών αρχών σε τέτοιου είδους διεργασίες. Θέλω να επιβεβαιώσω ότι δεν δεχόμεθα ατομικά παράπονα σε σχέση με την Λευκορωσία διότι οποτεδήποτε υπάρχουν θέματα με μια τρίτη χώρα ε, δεν διστάζει κανείς ή δεν θα έπρεπε να διστάζει να αναφέρεται σε εμά για τέτοιου είδους παρατυπίες. Κατά τα τελευταία έτη είχαμε ε, ε, επανειλημμένα τέτοιου είδους ε, δράσεις. Τίποτα λοιπόν δεν επιβεβαιώνει ότι υπάρχει εδώ συστηματική παραβίαση με τα όσα ισχυρίζεται ο αναφέρον ευρωπαϊκού δικαίου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ερωτώ τώρα τους συναδέφους ε, αν θέλουν να παρέμβουν για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχουν σοβαρές κατηγορίες που γύρονται από τον κύριο Σούμαρ. Τώρα ακούσαμε ότι αυτές οι κατηγορίες είναι αβάσιμες. Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι αβάσιμοι και υπήρξαν στοιχεία σε σχέση με στοιχεία που δεν υπάρχουν για να ε, τις αποδεικνύουν τις κατηγορίες αυτές και σε σχέση με τα όσα αναφέρθηκαν από τις πολωνικές αρχές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το θέμα αυτό εξετάστηκε σε βάθος και επαρκώς και τέτοιου είδους εγκληματικές δραστηριότητες σε σχέση με το πολωνικό ε, σύστημα δεν ε, υφίστανται. Ένα πρόβλημα όμως ε, παραμένει και το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Είναι το πρόβλημα των μη επαρκών προξενικών στελεχών στις υπηρεσίες και που πρέπει από τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπιστεί. Όσον αφορά για παράδειγμα το Μίνσκ όμως δεν, είναι, δεν έχουν την πρόθεση να δώσουν τη δυνατότητα να αναβαθμιστούν ή να μπορέσουν να αυξηθούν τα στελέχη της πολωνικής υπηρεσίας στο Μίνσκ ώστε να μπορέσει το πρόβλημα να διευθετηθεί. Αυτό πρέπει να αναφερθεί διότι είναι κάτι επί του οποίου δεν είναι δυνατόν εμείς να ασκήσουμε την επιρροή Άρα λοιπόν παρακαλώ νομίζω ότι πρέπει να κλείσει η αναφορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Εσείς παρακαλώ έχετε τον λόγο και σε σχέση με την ε, εκπόνηση αυτών των ε, θεμάτων από πλευράς Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών η θέση μας στο Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με τα ζητήματα αυτά ήταν ότι μπορεί ίσως να μην είναι κάτι μόνιμο αυτό, ωστόσο όμως αφορά το θέμα του outsourcing και γι' αυτό από πλευράς της ε, Επιτροπής που ίσως θα μπορούσε να ε, λάβει υπόψη τα θέματα αυτά σε σχέση με την πολωνική πρεσβεία. Γίνεται χρήση της διαδικασίας outsourcing και σε σχέση με την ε, διακρύβωση αυτή ε, όταν τίθεται ένα αίτημα για χορήγηση θεώρησης διαβατηρίου στην συνέχεια ο προξενικός κόμβος που δημιουργήθηκε για αυτή την ε, διαμεσολάβηση είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μας κάνει να δούμε πώς προχωρούν τα πράγματα στη Λευκορωσία για την ε, προώθηση ενός τέτοιου αιτήματο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για αυτό το θέμα. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν αντίστοιχα υπηρεσίες σε διάφορα σημεία για παράδειγμα, λειτουργούν οι υπηρεσίες αυτές από την 1η Νοεμβρίου και υπήρξαν σε σχέση με τις προξενικές υπηρεσίες οι ε, ενδείξεις ότι μπορούν οι ετούντες να θέσουν άμεσα το αίτημά τους στην αντίστοιχη υπηρεσία και μετά να τύχουν ανταπόκρισης στο αίτημά τους αυτό. Ευχαριστώ. Just, I join my colleagues also in proposal to close the petition and we see that... Παρακαλώ. Υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτές τις ε, θεωρήσεις ε, στη Λευκορωσία, αλλά παρόλα αυτά από τα στοιχεία που έχουμε λάβει δεν εκτιμούμε ότι πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Σούμαρ. Κύριε Σούμαρ, το πρόβλημα είναι το εξή. Το θέμα που θέτετε εδώ Το θέμα που θέτεται είναι ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή κατηγορία, ένας πολύ σοβαρός ισχυρισμός για υπαλλήλου και, και της πολωνικής δημοκρατίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχετε κάποια απόδειξη κύριε Σουμάρ. Και οποιοδήποτε δικαστήριο στον πλανήτη θα σας, ε, θα σας έκανε την ίδια α, ερώτηση. Εγώ είμαι Σλοβάκος. Έχω ζήσει υποκομμουνιστική δικτατορία επί 35 χρόνια. Φαντάζομαι λοιπόν πολύ καλά τι μπορεί να συμβαίνει σε μια κοινωνία σαν τη Λευκορωσική. Αλλά οφείλω να σας θέσω αυτήν την ερώτηση. Και καταλαβαίνω βεβαίως ότι η Λευκορωσία είναι σε μια δύσκολη θέση, ε, είναι σε μια διαδικασία εκδημοκρατισμού. Ε, έχω κατανόηση για τους Λευκορώσους πολίτες ε, και πιστεύω ότι η Λευκορωσία ανήκει στην Ευρώπη, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ. Έχετε αποδείξει για αυτά που λέτε. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες επιρροές από κάποια οργάνωση κτλ. Ε, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε σίγουροι ότι οι υπάλληλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης δουλεύουν με τίμιο και ξεκάθαρο τρόπο. Και για να σας πάρουμε στα σοβαρά χρειαζόμαστε κάποιες αποδείξεις. Αν υπάρχει περίπτωση διαφθοράς θα πρέπει κάπως να αποδειχθεί. Και εγώ πιστεύω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που λέει ότι έκανε το καταδύναμη για να ε, εξετάσει το πρόβλημα αυτό. Η Πολωνία έκανε ό,τι μπορούσε για να δει τι πρόβλημα υπήρχε με αυτές τις θεωρήσεις. Εσείς έχετε κάποια στοιχεία να μας δώσετε. Σας δίνω ξανά το λόγο. Είμαι επίκος τρίτης χώρας και μπορώ να ακούσω διάφορα εγώ όμως εφιστώ την προσοχή σας στις ε, πολλαπλές δηλώσεις ε, πολωνών ε, αξιωματούχων. Του εκπρέσβη για παράδειγμα της Πολωνίας στη Λευκορωσία. Συγκεκριμένα η πρέσβης που στον τύπο ανέφερε ότι στη Λευκορωσία εγκληματική συμμορία ελέγχει αυτή την επιχείρηση χορήγησης θεωρήσεων Σέγγεν και ελέγχει, είναι ένα κύκλωμα που ελέγχει το σύστημα αυτό. Θα σας παρακαλούσα να μου απαντήσετε. Τι γίνεται με την πολιτική της Γαλλίας, της ε, Δανίας, της Γερμανίας, της Ισπανίας. Πώς να το πω. Πρόκειται για πολλαπλές ε, παραβιάσεις ό,τι αφορά τη χορήγηση ε, θεωρήσεων το 2011. Που έγινε και σκάνδαλο. Τι έγινε μετά. Ο διευθυντής, ο υπεύθυνο ε, του πολωνικού προξενείου, που είχε ε, παράνομη θεώρηση Σέγγεν, μετατέθηκε και πού πήγε στη Λευκορωσία, στη χώρα μου. Ε, λυπούμε που δεν μπορώ να εκφραστώ όπως θα ήθελα γιατί είμαι πολύ νευρικός. Ε, Τέλος πάντων, αφού έφτασε λοιπόν στη χώρα μου, ξεκίνησε αυτή η ίδια ε, δουλειά, η ίδια επιχείρηση. Νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε πληροφορίες από τις τέσσερις αυτές χώρες. Τι έγινε το 2011 εκεί. Και αυτό που λέει η Κομισιόν ε, έρχεται σε αντίφαση, φάσκη και αντιφάσκη Κομισιόν, η οποία είχε παραδεχθεί ότι υπήρξαν δυσκολίες ε, σε ό,τι αφορά την χορήγηση θεωρήσεων Σέγγεν στη Λευκορωσία. Σε μία δε από τις επιστολές της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συμβουλεύει να μην πάω σε κάποιον νομικό μεσολαβητή, λέει ο μιλητής. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα όμως. Δεν επιλύεται έτσι το θέμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εκπρόσωπο της πολωνικής πλευράς, την εκπρόσωπο, συγγνώμη, της πολιτικής πλευράς, είπε πως το Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας έλεγξε επανειλημμένως τα διάφορα προξενέα της Πολωνίας στη Λευκορωσία. Όμως, This, uh, I think δεν μπορούμε να πιστέψουμε τα πορίσματα αυτού του ελέγχου. Γιατί ουσιαστικά οι ελέγχοντες ε, ήταν οι ελεγχόμενοι ταυτόχρονα. Τώρα σε ό,τι αφορά τις αποδείξεις γιατί μου ζητήσατε να σας ε, προσκομίσω αποδείξεις. Εγώ ευχαρίστως να σας δώσω όλα τα έγγραφα, όλες τις πληροφορίες. Έχω και μάρτυρες, αλλά δεν μπορούν να έρθουν εδώ γιατί είναι κάτοικοι και οι πίκοες δεν μπορούν να έρθουν εδώ. Αυτή η αναφορά που αφορά τη Λευκορωσία εξετάζεται εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά ο τύπος, ε, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωση στη Λευκορωσία δεν έχει πει κουβέντα για αυτό το θέμα. Διότι το ελέγχουν, ε, ελέγχεται η κατάσταση από το λευκορωσικό καθεστώς που αποκομίζει κέρδος από όλη αυτή την ε, επιχείρηση. Και όταν υπήρχε αυτό το κύκλωμα για την παράνομη έκδοση θεωρήσεων Σέγγεν, ήρθε, ε, ήρθαν κάποια μέτρα σε ό,τι αφορά τη, το χώρο Σέγγεν και όταν ήρθα εγώ εδώ μου δόθηκαν πέντε λεπτά στην Επιτροπή σας για να παρουσιάσω αυτή την υπόθεση. Όμως είναι πάρα πολύ σοβαρή. Σας το είπα και πριν η κατάσταση. Και θα ήθελα να σας δώσω πιο αναλυτικές πληροφορίες. Απλά θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε λίγο περισσότερο χρόνο. Ή ίσως μια ακόμη δυνατότητα να παραστώ εδώ και να σας δώσω όλα αυτά τα στοιχεία. Στην πραγματικότητα, δεν σας έδωσα αποδείξεις. Έχετε δίκιο. Απλά δεν μπορούσα να το κάνω σήμερα. Απλά λοιπόν σας παρακαλώ να μου δώσετε αυτή τη δυνατότητα να το κάνω σε κάποια άλλη ε, ευκαιρία. Να σας δώσω δηλαδή αποδεικτικά στοιχεία για αυτή την υπόθεση. Ο Πρόεδρος. Κύριε Σουμάρ, δεν θα σταματήσει εδώ ε, όρους της ιστορίας. Στο μέλλον φυσικά και μπορείτε να λάβετε οποιοδήποτε μέτρο θεωρήσετε εσείς σόφρον και να κάνετε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρείτε σκόπιμη. Απλά Έχουμε ακολουθήσει όλα τα βήματα αυτής της διαδικασίας. Ε, πολύ ενδελεχώς ερευνήσαμε ε, όλο το φάκελο. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχω λάβει εγώ ή εμείς κανένα, ούτε ένα αποδεικτικό στοιχείο ή έγγραφο που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το οποίο να αποδεικνύει ότι εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ε, ένα κρούσμα διαφθοράς ή κρούσματα διαφθοράς. Γι' αυτό λοιπόν ε, και αστρέφω στους συναδέλφους, επειδή δεν έχουμε λάβει αποδεικτικά στοιχεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ερευνήσει το θέμα σε βάθος, όπως και η Πολωνία, προτείνω τρία πράγματα για σήμερα. Πρώτον, θα ήταν λογικό πιστεύω και σόφρον να, γράψουμε μια επιστολή στη λευκορωσική κυβέρνηση και να την προειδοποιούμε ότι έχουμε λάβει αυτά τα στοιχεία, αυτές τις πληροφορίες και να εφιστούμε την προσοχή του στο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επανεξετάσει το σύστημα έκδοσης θεωρήσεων και θα εφαρμόσει μια πολύ πιο αυστηρή διαδικασία και θα ήθελε να υπάρχει και η συνεργασία από πλευρά της Λευκορωσίας. Θα γράψουμε επίσης επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία θα ενημερώνουμε την Κομισιόν ότι με βάση τις προφορές που λάβαμε ζητούμε η Κομισιόν να εξετάσει το ζήτημα το οποίο εσείς κύριε αναφέροντα εγείρατε. Ότι δηλαδή με εξωτερική ανάθεση ενδεχομένω με τέτοιε διαδικασίες, θα μπορούσε ενδεχομένω να προκύψει αυτή η περίπτωση, δηλαδή να εκδοθεί μία ευρωπαϊκή βίζα και να δοθεί ε, με παράνομα θέμητο τρόπο ή μη ορθό τρόπο σε πολίτη της Λευκορωσίας. Πάντως, συγκεκριμένες αποδείξεις δεν έχουμε λάβει μέχρι σήμερα. Εγώ λοιπόν προτείνω να κλείσει αυτή η αναφορά και να προσθέσουμε ότι στο μέλλον μπορείτε εσείς να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρείτε σκόπιμη ή ενδεδειγμένη. Αλλά προς το παρόν δεν βλέπω κανένα στοιχείο, καμία απόδειξη, καμία γνωμοδότηση ή οτιδήποτε άλλο βάσει του οποίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσε να λάβει οποιοδήποτε μέτρο. Καθιουδήποτε προσώπου, εξωματούχου ή άλλου. Και ρωτώ αν συμφωνούν οι συναδελφοί μου. Μάλιστα, συμφωνούν. Σας ευχαριστώ πολύ κυρίε και κύριοι. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνω τη σημερινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Καλό απόγευμα, καλό βράδυ. Θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί.